Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Ρόμπερτ Άτκινς δεν, δεν είναι πλέον μέλος της Επιτροπής Μεταφορών. Η διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίασή της 8 Ιανουαρίου 2009 και σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού 45